Το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η σύντομη παρουσίαση των ακόλουτων εκθέσεων. Ε, κυρία Ροζιέ, θεμητά μέτρα για την προστασία των καταγγελόντων που ενεργούν προς το δημόσιο συμφέρον. Ε, το λόγο έχει η συγγήτρια για τέσσερα λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Όταν παρουσιάζει κανείς μια τέτοια εργασία, ευχαριστεί τους συναδέλφους για τη συνεργασία. Θα το έκανε ευχαρίστω, αλλά προτιμώ να ευχαριστήσω πρώτο, τον κύριο Δελτούρ, την κυρία Αλέ, τον κύριο, την κυρία Φρασόν, όλους αυτούς που μια μέρα έκαναν αυτή τη γενναία επιλογή, την τολμηρή επιλογή να μιλήσουν. Δεν είναι εύκολο, γιατί οι καταγγέλλοντες, κάνουν αυτήν την επιλογή της εντιμότητας, της αλήθειας, της ε, και με κίνδυνο πολλές φορές της ίδιας της ζωής τους. Ε, είναι η πρώτη φορά που το Κοινοβούλιο εγκρίνει ένα κείμενο για την προστασία των καταγγελόντων και είναι αρκετά εκπληκτικό γιατί οι αποφάσεις έχουν αναλυθεί ήδη στο επίπεδο άλλων θεσμικών οργάνων όπως το Συμβουλίο που από το 2014 έχει εγκρίνει μια απόφαση με στόχους φιλόδοξους και αρκετά ε, αποτελεσματικούς φαίνεται. Σε αυτούς βασιστήκαμε σε μεγάλο βαθμό. Ε, ευχαριστώ λοιπόν όλους τους καταγγέλλοντες. Τώρα να πω ότι το Κοινοβούλιο κάλεσε πολλές φορές την προστασία των καταγγελόντων στο επίπεδο ψηφίσματος, ε, κυρίως μετά το, ε, την υπόθεση LuxLeaks και την, ε, το έργο της Επιτροπής TAX 1 και TAX 2. Ε, τιμήσαμε βεβαίω ε, για να με το ε, βραβείο των Ευρωπαίων Πολιτών. πολλά πετύχαμε χάρη σε αυτού του καταγγέλλοντε, αλλά σήμερα ο Αντουάν Μπερτούρ και η κυρία Δέλα έχουν καταδικαστεί σε φυλάκιση με αναστολή. Παρακολουθούμε την καθημερινότητα των Ευρωπολιτών. Θέλουμε να ε, υπάρξει καταπολέμηση φοροδιαφυγή, όμω αυτοί οι άνθρωποι, με όσα προσέφεραν, είναι καταδικασμένοι. Θέλουμε λοιπόν σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο, ε, καλείται σήμερα το Ευρωκοινοβούλιο, να εγκρίνει ένα εργαλείο για την προστασία των καταναλώντων σε όλη την Ευρώπη. Αυτό το κείμενο μπορεί να αποτελέσει το θεμέλιο για μια αποτελεσματική προστασία. Όλο ιδιαίτερο προτείνουμε μια, έναν ευρύ ορισμό για του ε, καταγγέλλοντε είτε είναι σύμβουλοι, μισθωτοί, ε, εξωτερικοί συνεργάτες. Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Μας ενδιαφέρει το είδος της πληροφορίας που καταγγέλλεται. Από τη στιγμή λοιπόν που ένας καταγγέλων ε, εντοπίζει ε, δράσεις ή κινήσεις που αντίκεινται στο ευρωπαϊκό ένομο συμφέρον, αυτό μπορεί να θεωρηθεί καταγγελία με την έννοια του καταγγέλλοντος πολλές φορές δέχονται τεράστιες πιέσεις αυτοί οι άνθρωποι. Πολλές φορές απειλούνται με αντίπεινα. Αυτά τα αντίπεινα πρέπει να είναι αξιόπινα και πρέπει να τιμωρούνται. Και η ζημία που προκαλείται στον καταγγέλλοντα και τον περίγυρό τους πρέπει να ε, είναι αντικείμενο αποζημίωσης. Θα πρέπει οι καταγγέλλοντες να ε, λάβουν δικαστική συνδρομή, οικονομική ηθικού χαρακτήρα, διότι πολλές φορές ε, χάνουν τη δουλειά τους, ε, οι συνθήκες διαβίωσης τους χάνονται, χάνουν το σπίτι τους, ε, χάνουν τους πόρους τους. Χρειάζεται πολλές φορές λοιπόν οικονομική υποστήριξη αλλά και ψυχολογική υποστήριξη διότι οι άνθρωποι αυτοί έρχονται αντιμέτωποι με οργανισμούς που έχουν τεράστια μέσα και πίεσης και πειθούς. Θα πρέπει λοιπόν εδώ οι άνθρωποι αυτοί, εφόσον είναι μισθωτοί, ε, σε μια εταιρεία να αναλυφθούν τα απαραίτητα μέτρα ώστε ο εργοδότης του να μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα χάσει τη δουλειά του λόγου χάρη. Θα πρέπει να προβλέψουμε ανεξάρτητες αρχές για να υποδεχτούν, να βοηθήσουν και να ε, υποστηρίξουν, να συμβουλεύσουν τους καταγγέλλοντες. Ε, πολλές φορές, όπως είπα, έρχονται αντιμετώπιοι με ισχυρούς οργανισμούς οι άνθρωποι αυτοί. Η ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αρχή που θα μπορούσε να ε, είναι ε, υπεύθυνη για τον συντονισμό και να είναι και μια δίωδος προσφυγής για τους καταγγέλλοντες θα ήταν σημαντικό. Ένα άλλο σημαντικό πλαίσιο που θα συζητήσουμε αυτή την εβδομάδα, άλλου χαρακτήρα, είναι όλα αυτά τα άτομα που έχουν πέσει θύματα της γλυφωσάτης. Εδώ υπήρξε καταγγελία κατά της Μονσάντο, υπήρξε καταγγελία στις εθνικές αρχές. Ε, δεν ε, ακούστηκε όμως, θα ήταν σημαντικό να υπήρχε ανεξάρτητη Ευρωπαϊκή Αρχή για τις καταγγελίες λόγου χάρη. Αλλά να καταγγείλω και ε, μία πρακτική αρκετά ε, καταδικαστέα κάποιων ε, μελών του ημικυκλίου. Κάποιοι θέλουν τους καταγγέλλοντες, αλλά δεν θέλουν να έχουν οι καταγγέλλοντες κανία δυνατότητα να έχουν πρόσβαση στον τύπο. Μα στις σοβαρότερες υποθέσεις, στις σοβαρότατες ε, παραβιάσεις, με ε, καταχρήσεις και υπεξαιρέσεις, με διαφθορά. Ε, πώς δεν θα πάνε στον τύπο οι καταγγέλλοντες. Είναι πλέον εκτεθειμένοι τι νόημα θα είχε να καταργηθεί η προστασία τους για τις σοβαρότατες ακριβώς υποθέσεις όπου θα έπρεπε σημειωτό, σημειωτό, κατευθείαν μάλλον να βρεθούν ε, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης καταγγελίες τους. Είναι λοιπόν ε, νομίζω ε, πραγματικά κρίμα αύριο που θα αποτίσουμε φορό τιμής στην κυρία Καρουάνα Γκαλίτσια να ε, μην ψηφίσουμε υπέρ μια τέτοια προστασία. Ελπίζω να το δείξουν όλοι αύριο στην αυριανή ψηφοφορία. Σα ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ροζιέρ. Και τώρα η διαδικασία ΚΑΤΣΤΙΑΗ. Η κυρία Σόιντροβα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε ένα νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των καταγγελόντων, ειδικά σε, εθνικό σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι άνθρωποι αυτοί, οι καταγγέλλοντε, που αποφασίζουν να αποκαλύψουν εμπιστευτικέ πληροφορίε, απόρριτε πληροφορίε για παράνομε δραστηριότητε, που βοηθούν στην καταπολέμηση τη απάτη, τη διαφθορά, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή. Λογικό είναι να προστατεύονται βεβαίω. Όταν προτείνουμε έναν ευρωπαϊκό κανονισμό, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, διότι όταν μιλάμε για ανωνυμία, δεν είναι το ίδιο με την εμπιστευτικότητα κάποιοι. Πρέπει να γνωρίζουν την ταυτότητα των ατόμων αυτών. Όμω, καλύτερα να είναι γνωστοί στι αρχέ ε, επίβλεψη, στι αρχέ υποπτία. Πρέπει λοιπόν να προστατεύσουμε του ε, καταγγέλλοντε, αλλά να είμαστε βέβαιοι ότι τους προστατεύουμε αναλόγω με τα όσα μας προσφέρουν με τις καταγγελίες τους. Δηλαδή το δικαίωμα στην προστασία των καταγγελόντων είναι σημαντικό, αλλά στο ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασίας πρέπει να σκεφτούμε και τα εθνικά πλαίσια που υπάρχουν και να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κυρία Γουόρτ. Οι καταγγέλλοντε είναι με ύψη τη σημασία για την προστασία του δημόσιου συμφέροντο, για την προστασία των δημοσίου, του δημοσίου χρήματο, για τη διαφάνεια και την ακαιρεότητα του δημόσιου πολιτικού βίου. Υπό το φω των πρόσφατων σκανδάλων και όλο ιδιαίτερω μετά την τελευταία, την δολοφονία τη τελευταία εβδομάδα τη Μαλτέζα δημοσιογράφου Δάφνη Καρουάνα Γκαλίτσια. Είναι σημαντικό να έχουμε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο προστασία. Για την προστασία των καταγγελόντων πρέπει να σκεφτούμε την προστασία των δημοσιογράφων και των πηγών του, την προστασία των μη κυβερνητικών οργανώσεων, την ελευθεροτυπία και την αλήθεια που προστατεύουμε μαζί. Ε, η ομάδα μου έχει ε, διδραματίσει σημαντικό ρόλο στην πρόθεση τη ευρωπαϊκή δράση για την προστασία των καταγγελόντων και θέλω να ευχαριστήσω την συνάδελφο Βυριζινή Ροζιέρη για τη δουλειά τη για την έκθεση αυτή. Η διαφάνεια, η δημοκρατία, η ελευθεροτυπία, τα υψηλά ε, διοντολογικά πρότυπα και προδιαγραφέ σε δημόσιου και ιδιωτικού φορεί, αυτά είναι οι αρχέ που θα προστατεύσουμε προστατεύοντα του καταγγέλλοντε. Πρέπει λοιπόν να παραμείνουμε είναι ε, άφοβα και χωρίς να διστάσουμε όταν άλλες ομάδες δεν θέλουν την ίδια προστασία απέναντι ε, στους όσους έχουν αντιρρήσεις, όπως το ΕΛΚ κυρίως. Πρέπει να ε, υποστηρίξουμε την διαφάνεια και όχι να κλείσουμε την πόρτα ή να τραβήξουμε τις κουρτίνες για να μην βλέπει ο κόσμος. Ευχαριστούμε κύριο κύριος Μαριάς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σε μια φάση όπου πραγματικά η ευρώπη έχει εκατομμύρια ανέργους όπου έχουμε εκατομμύρια φτωχούς και ταυτόχρονα τεράστιο δημόσιο χρέος είναι βέβαιο ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με αποφασιστικότητα η φοροδιαφυγή η φοροαποφυγή και φυσικά η διαφθορά. και στην πάλη αυτή σε αυτόν τον αγώνα σημαντικό ρόλο παίζουν οι καταγγέλλοντες οι οποίοι είτε εργάζονται στο δημόσιο είτε στο ιδιωτικό τομέα και οι οποίοι αποκαλύπτουν πραγματικά τα σκάνδαλα τα οποία συμβαίνουν πρέπει λοιπόν να υπάρξει μια προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και επίσης να δοθεί η δυνατότητα να μπορούν να προσέρχονται αυθορμήτως αλλά αν ξέρουν ότι θα τιμωρηθούν προφανώς θα είναι πολύ δύσκολο να έχουμε τους καταγγέλλοντες. είναι σημαντικό ότι είχαμε τη λίστα φαλτσιάνη αυτό που ονομάζεται στην ελλάδα λίστα λαγκάρτ που αποκάλυψε τεράστια φοροδιαφυγή η οποία έχει συμβεί και στην ελλάδα. προστασία λοιπόν των καταγγελλόντων χάρη του δημοσίου συμφέροντος και γι' αυτό θα πρέπει να υιοθετήσουμε ένα ευρύ ορισμό της έννοιας του καταγγέλλοντος να λαμβάνουμε υπόψη κυρίως το είδος της πληροφορίας και φυσικά να υπάρχει και προστασία τους ακόμη και οικονομική στήριξη αν θέλουμε πραγματικά οι καταγγέλλοντες να προσέρχονται και να αποκαλύπτουν αυτά τα οποία συμβαίνουν σε βάρος του δημοσίου συμφέροντος. ευχαριστώ. Επόμενος, ε, Κύριε Πρόεδρε, οι καταγγέλλοντες είναι απαραίτητοι και γι' αυτό πρέπει να τους προστατεύουμε. Θα ήθελα λοιπόν να ευχαριστήσω τον, ε, την εισηγήτρια για αυτό το εξαίρετο έγγραφο. Ε, είχε έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Έπρεπε πια να υπάρχει το έγγραφο αυτό. Όταν μιλάμε για ελευθερία και δημοκρατία, ε, συνήθως ε, είμαστε στην αιχμή του δώρατος. Εδώ όμως είχαμε καθυστερήσει πάρα πολύ. Και θυμάμαι κάποια παραδείγματα από την Κροατία. Εκεί έχουμε ένα πολύ γνωστό παράδειγμα ενός ε, καταγγέλλοντος ε, στην πετρελοβιομηχανία, στην εταιρεία Ίνα της Κροατίας. Ήταν δημόσια υπάλληλος, δούλευε για το δημόσιο. Ε, εγώ Θεωρώ ότι το Κοινοβούλιο πρέπει να στηρίζει αυτούς οι οποίοι ε, έχουν στόχο να πράξουν κάτι καλό. Και τώρα... Κύριε Φάρμαγκαν, παρακαλώ. Όταν μιλάμε για καταγγέλλοντες, ακούγονται πολλά μεγάλα λόγια. Όλοι λένε ότι είναι σημαντικοί, είναι θαραλέοι, είναι μοναδικοί αλλά μόνο αν τελικά μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια κατάσταση όπου οι άνθρωποι δεν θα πρέπει να είναι θαραλέοι για να καταγγείλουν κάτι. Θα είναι φυσιολογικό να καταγγέλει κανεί το κακό. Μόνο τότε θα έχουμε πετύχει, γιατί αυτή τη στιγμή πρέπει κανεί να είναι η εξαίρεση. Γιατί στη δική μου τουλάχιστον τη χώρα, αν καταγγείλει κανεί κάτι, ε, τελικά ε, θα καταλήξει στο να είναι άνεργος, ε, να καταστραφεί πνευματικά, ψυχολογικά. Και το έχω βιώσει συμβεί αυτό πάρα πολλές φορές. Στη δική μου τη χώρα έχω βιώσει καταστάσεις ε, όπου είχαν υπάρξει ακόμα και ε, ψεύτικες ε, αιτιάσεις εις βάρους τους ε, ότι ήταν παιδόφιλοι ενώ δεν ήταν απλά και μόνο επειδή είχαν καταγγείλει. Τους βάλανε και ποντίκια. Ε, τραγικά πράγματα. Πρέπει λοιπόν να τους βοηθήσουμε. Δεν μπορούμε να τους λέμε μη μιλάτε γιατί κινδυνεύει η ζωή σας. Ελπίζω αυτή η κατάσταση να αλλάξει. Και θέλω να πιστεύω αυτό ήταν μια καλή αρχή. Ο κύριος Καπούτο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια οι καταγγέλλοντες διδραματίζουν σημαντικό ρόλο στο να αποκαλύπτουν ε, παραβιάσεις ε, νομοθεσίας ε, και υπήρξε και μια σειρά ολόκληρων σκανδάλων σε πάρα πολλούς τομείς. Η προστασία της δημόσιας υγείας, το περιβάλλον, στην φοροδιαφυγή. Αυτή λοιπόν η καταγγελία είναι ένα πολύ σημαντικό εργαλείο προς όφελος του κοινού συμφέροντος. Δυστυχώ, βέβαια δεν υπάρχει ουσιαστική προστασία και δεν μπορούμε να αγγιητούμε και ένα αποτελεσματικό πλαίσιο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουν υπάρξει πολλοί διεθνείς κανόνες για να προστατεύονται οι καταγγέλλοντες. Ως εκ τούτου θα πρέπει σε αυτά να βασιστούμε ως Ευρώπη. Και με βάση αυτούς τους κανόνες ο ορισμός του καταγγέλλοντος θα πρέπει να είναι αρκετά ευρύς, να καλύπτει όσο δυνατόν περισσότερες καταστάσεις και να προστατεύει με ανεξάρτητο τρόπο και τον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Και τους ε, συμβούλους ε, και τους ελεύθερους επαγγελματίες Έχουμε την περίπτωση της κυρίας Γκαλίτσια, η οποία ορίστηκε ως η γυναίκα των Wikileaks. Εμείς βέβαια θα πρέπει παρόλα αυτά να προσπαθήσουμε να προστατεύουμε τους καταγγέλνους και να τους βγάλουμε από λάθος, από τη σκιά που έχει πέσει τώρα στο συνδυότητά τους. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ο Επίτροπος Μοσκοβιξή είπε την ε, περασμένη εβδομάδα ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι πρωτοπόρο στην καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του ξεπλήματος χρήματος. Χωρίς τη δουλειά του κυρίου Ντελτούρ δεν θα μπορούσαμε να το είχαμε πετύχει. Είναι ο καταγγέλων από το Λουξεμβούργο που ευθύνεται που χάρη σε αυτόν, ε, σε χρωστάμε τα LuxLeaks, τα Η κυρία Γκαλίτσια είχε έρθει και είχε δώσει πληροφορίες στην Επιτροπή μας για τις φορολογικές υποθέσεις των πλούσιων στη Μάλτα. Αυτοί οι δύο θαραλέοι άνθρωποι μας έδωσαν τις πληροφορίες που χρειαζόμαστε για να καταγγείλουμε και να αποκαλύψουμε την συμπεριφορά της ευρωπαϊκής πλουτοκρατίας. Ε, οι λαοί όλο και περισσότερο χάνουν την εμπιστοσύνη τους στο σύστημα η μία δολοφονήθηκε και ο ένας ε, και ο άλλος, ο κύριος Δελτούρ, ε, καταδικάστηκε. Ενώ αυτοί μας είχαν καταγγείλει και μας είχαν αποκαλύψει αλήθειες. Πώς η διαφθορά παραμένει κρυφή, γιατί όσοι τη γνωρίζουν φοβούνται να παρουσιαστούν. Αναρωτιέμαι. Η νομοθεσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έτσι όπως προτείνεται, δίνει την προστασία στους καταγγέλλοντες ε, την οποία χρειάζονται. Ευχαριστούμε την κυρία Σκοτ Κάτω και τώρα η κυρία Κατρίνα Κινίτσι έχει το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Οι αποκαλύψεις του Panama Papers, του LuxLeaks ε, και ούτω καθεξής είναι ε, μεγάλα σκάνδαλα που αποκαλύφθηκαν και έδειξαν υποθέσεις διαφθοράς και φοροαπάτης απάτης, με την τολμηρή πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων ε, που αποφάσισαν να καταγγείλουν δράσεις που έβλαπταν το σύνολο των πολιτών. Το Κοινοβούλιο καλώ λοιπόν λαμβάνει μέρη για ένα θέμα τόσο ευαίσθητο και επίκαιρο, γιατί υπάρχει διαφορά στα νομοθετικά συστήματα των κατώμελων σε όσα προβλέπουν για την προστασία των καταγγελόντων, οι οποίοι δεν θα προστατεύονται καν ή πολλέ φορέ και ποινικοποιούνται για την, ε, οι δράσει του, οι αποκαλύψει του. Ευχαριστώ λοιπόν την εισηγήτρια για τη δουλειά τη, γιατί έδειξε πόσο απαραίτητο είναι ένα αριθμιστικό πλαίσιο που να προβλέψει ελάχιστε προδιαγραφέ για να εναρμονίσουμε την ε, εξέταση υποθέσεων και να προστατεύσουμε του ε, αδειοδότε, του καταγγέλλοντε, με συγκεκριμένε νομικέ ρυθμίσει, αναγνωρίζοντα το θεμελιώδη ρόλο του στο δημόσιο πολιτικό βίο. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κινίτση. Ο κύριος Φάμπιο Μάσιμο Καστάλντο έχει το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Μιλάμε για προστασία των whistleblowers, των καταγγελόντων και μιλάμε και για πραγματική ε, διαφάνεια, για πραγματική καταπολέμηση της διαφθοράς. Όμως, πέρα από τα λόγια, ε, τα στοιχεία μας δείχνουν ένα τελείως διαφορετικό νομοθετικό σύστημα από χώρα σε χώρα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή υπάρχουν χώρες που έχουν ε, προβλέψει συστήματα στο ύψο των περιστάσεων, ενώ άλλα επιτρέπουν, επιβάλλονται και ποινέ. Πρέπει λοιπόν να υπάρξει ουσιαστική δράση, όχι μόνο ε, θεωρητική. Θα πρέπει οι καταγγέλλοντε ανώνυμοι να μπορούν να αποκαλύπτουν και να του ε, προστατεύουμε από του εργοδότε του, από του οργανισμού για του οποίου εργάζονται. Αυτό, κατά τη δική μου την άποψη, είναι σημαντικό πριν να υπάρξει αντιστροφή του βάρου απόδειξη. Σε περίπτωση συμπεριφορών δράσεων ε, που μπορεί να είναι συνώνυμα με διακριτική μεταχείριση, θα πρέπει τις αποδείξεις να μην πρέπει να τις ε, παρέχει ο, παρά μόνον ο καταγγέλων που θα δείχνει ότι έχει υποστεί ζημιά με οικονομικές συνέπειες. Αυτό πρέπει πραγματικά να κάνουμε αν θέλουμε να μιλάμε για προστασία των καταγγελόντων. Ιδάλλως για το θάρρος τους με τα λόγια το μόνο που θα πετύχουμε είναι να παρατείνουμε τη σιωπή μας και την αδιαφορία μας. Ευχαριστούμε κύριε Καστάλντο. Τελευταίος και εξίσου σημαντικός Τελευταία και εξίσου σημαντική, κυρία Ρουοχόνεν λένε. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε, συγκλονιστήκαμε όλοι με τη δολοφονία πριν από λίγες μέρες της ε, τολμηρής δημοσιογράφου της Θαραλέας Δάφνης Γκαλιτσιάνα η οποία αποκάλυψε περιπτώσεις υπεξαίρεσης χρημάτων, διαφθοράς και τέτοιου είδους φορολογικών και άλλων ε, αδικημάτων. Είναι παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί στους καταγγέλλοντες, στους whistleblowers και πώς πρέπει να προστατεύονται. Έχουμε τις, τους διάβλους, τις διάβλους ε, ανώνυμης κοινοποίηση και γνωστοποίησης. Υπάρχουν καλά πράγματα λοιπόν μέσα σε αυτό το κείμενο και θα πρέπει να βοηθηθούν και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για να λειτουργήσουν καλύτερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειαζόμαστε σαφή ε, κανονισμό έτσι ώστε να ε, προστατεύσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους που καταγγέλουν τις υπεξερέξεις και τα δικήματα της επιχείρησης στην οποία εργάζονται. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος. Και εγώ σας ευχαριστώ. Τόμασιτς, παρακαλώ, κύριε Η κυρία Τόμασιτς. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ξέρετε, οι καταγγέλλοντες είναι πολύ σημαντικοί, οι whistleblowers, για όλες τις κοινωνίες, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι διακινδυνεύουν το δικό τους μέλλον, ε, γιατί θέλουν να προσπίσουν το δημόσιο συμφέρον και συχνά οι κοινωνίες δεν δείχνουν την αναγνώριση που τους οφείλουν και τους περιθωριοποιούν τελικά αυτούς τους ανθρώπους. Είναι απαραίτητο να τους προστατεύσουμε για να ενθαρρύνουμε τους πολίτες να έχουν πραγματική αγωγή του πολίτη, δηλαδή να αποκαλύψουν καλύπτουν πληροφορίες που είναι υπέρ του δημοσίου συμφέροντος και μάλιστα χωρίς κανένα δισταγμό. Αναφέρομαι κυρίως στην εθνική νομοθεσία, την οποία θα πρέπει να έχουν όλα τα κράτη-μέλη και να προβλέπεται απόλυτη προστασία των καταγγελόντων. Ε, δεν μπορεί κανείς να το νομοθετήσει αυτό και να γίνει με ένα μαγικό ραβδάκι επειδή το νομοθέτησε. Γιατί ε, εάν θέλουμε να σταματήσουμε την άλλη πλευρά σε ορισμένες ε, περιπτώσεις μπορεί να προστατεύουμε και ανθρώπους που τελικά είναι υπόλογοι. Αυτό είναι κάτι που θα πρέπει λοιπόν να το αποφασίσουν τα δικαστήρια. Ευχαριστώ. Ο κύριος Επιτίδιος παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Τόσο στο δημόσιο τομέα όσο και στις μεγάλες επιχειρήσεις υπάρχουν ορισμένα άτομα τα οποία εκμεταλλεύονται τη θέση τους και προβαίνουν σε παράνομες δραστηριότητες όπως ε, απάτες, φοροδιαφυγές παράνομο πλουτισμό και άλλες ατασταλίες δημιουργώντας έτσι και συντηρώντας την ε, γενικότερη μορφή διαφθορά. αντιδρώντας αυτήν την απαράδεκτη κατάσταση ορισμένοι έντιμοι πολίτες καταγγέλουν όποιες παράνομες δραστηριότητες υποπίπτουν στην αντίληψή τους. δυστυχώς πολλές φορές οι άνθρωποι αυτοί πέφτουν θύματα της εντιμότητα και του θάρρους τους διότι διώκονται από τις εργασίε του, απειλείται η ζωή του, η ζωή των μελών τη οικογένεια του, πολλέ φορέ χάνουν και τη ζωή του και γενικώ υποφέρουν. επειδή με τι δραστηριότητε, αυτέ οι άνθρωποι αυτοί βοηθούν το κράτο να λειτουργήσει οφείλει το κράτο να του προστατεύσει και να μεθοδεύσει και να θεσμοθετήσει διαδικασίε οι οποίε θα συμβάλλουν στην ενίσχυση τη ε, προθυμία του να καταγγέλουν αυτέ τι παράνομε ενέργειε εδώ όμως πρέπει να προσέξουμε να μην υποθάλψουμε περιπτώσεις ψευδούς καταμηνύσεως και αντεκδικήσεως. δεν θέλουμε καταδότες θέλουμε ανθρώπους οι οποίοι θα καταγγέλουν παράνομες δραστηριότητες ούτως ώστε να λειτουργεί σωστά το κράτος με τις αρχές της χρυσής διοικήσεως και του κράτους δικαίου. ευχαριστώ πολύ. And now, on behalf Ευχαριστώ και τώρα εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ο Επίτροπος κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος έχει το λόγο. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στην εισηγήτρια για αυτή την έκθεση που αποτελεί σημαντική συμβολή στη συζήτησή μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ακράδαντα πεπισμένη ότι το να προστατεύει κανείς εκείνους που χτυπούν το σήμα του κινδύνου αυτό βοηθά να εντοπιστούν ουσιαστικές παραβάσεις του νόμου που αλλιώς δεν θα μπορούσαν να εντοπιστούν. Η καταγγελία είναι κάτι το ε, απολύτως απαραίτητο για να υπάρχει ουσιαστική επιβολή του νόμου και για να μπορούμε να διαπιλάξουμε το δημόσιο συμφέρον. Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω ότι οφείλουμε να προστατεύουμε την ε, υπεύθυνη καταγγελία που έχει ως στόχο και την προστασία του δημόσιου συμφέροντος. Είναι απολύτως απαραίτητο να διαφυλάσσουμε τα δικαιώματα και τα συμφέροντα ε, φορέων που επηρεάζονται από τις καταγγελίες, όπως ε, παραδείγματο χάνει το δικαίωμα της υπεράσπισης. Το θέμα είναι πώς μπορεί κανείς να επιτύχει αυτούς τους στόχους με τον καλύτερο τρόπο και πώς μπορούμε όλα αυτά να τα επιτύχουμε σε ενωσιακό επίπεδο. Όσοι γνωρίζετε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη στιγμή βρίσκεται στην τελική φάση ε, της διαμόρφωσης ε, της ε, δράσης της. Νομίζουμε ότι αυτό θα προκαλέσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λάβαμε περίπου 7.700 απαντήσεις, περίπου 200 εξ αυτών είναι από φορείς και θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι όσοι αντέδρασαν όλοι τάχτηκαν ανεπιφύλακτα υπέρ της προστασίας των καταγγελόντων. Όσον αφορά στους ε, τομείς με τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να προστατεύσει τα κράτη-μέλη και τους καταγγέλλοντες, η πρώτη τομείς είναι πρώτον στον αγώνα κατά της απάτης και της διαφθοράς. Κατόπιν, αγώνας ε, κατά της ε, φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής Επίσης, η προστασία του περιβάλλοντος και τέλος η προστασία της δημόσιας υγείας και ασφάλειας. Για να ολοκληρώσουμε την άποψή μας, αναθέσαμε μία μελέτη σε εξωτερικούς συνεργάτες για να χαρτογραφήσουμε την κατάσταση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπάρξουν στοχευμένες διαβουλεύσεις με εθνικούς φορείς και άλλους άμεσα ενδιαφερόμενους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά το πρώτο κομμάτι του 2018 θα συνεχίσει τις προσπαθειές της. Εδώ λοιπόν η έκθεσή σας είναι ιδιαίτερα επίκαιρη και ε, αυτά που προτείνατε θα τα λάβουμε υπόψη μας ε, στη δουλειά μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, ε, λέει ο Πρόεδρος, και ευχαριστούμε πολύ και κλείνω όλο